Okay. I will speak in... Θα μιλήσω ισπανικά. Use your headphones. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Okay. Bueno, la... Λοιπόν, ετήσια έκθεση το 2017 το Ευρωπαϊκό Ταμείου για τη Δημοκρατία από τον κύριο Τζέρσι Πομιανόφσκι. Θέλω να τον καλωσορίσω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία είναι πλήρως λειτουργικό από τον Ιούλιο του 2013 και ε, διαστηριοποιηθεί ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια της λειτουργία του, στηρίζοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει η ε, χρηματοδότηση και αποτελεί ένα σημαντικό ε, μέσο για τη στήριξη της δημοκρατίας. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών της και των κρατών μελών. Είναι όμως ένα ανεξάρτητο ίδρυμα ε, βελγικού δικαίου και η προστιθέμενη αξία του είναι ότι επιτρέπει να δοθεί μια γρήγορη χρηματοδότηση, σε λίγες μέρες δηλαδή, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει προβλήματα ή καθυστερήσεις ε, λόγω του ε, δημοσιονομικού μας κανονισμού. 380 πρωτοβουλίες έχει χρηματοδοτήσει μέχρι στιγμής από το 2015 και το γεωγραφικό πλαίσιο έχει διευρυνθεί πέρα από τις γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τους γείτονες των γειτόνων, όπως για παράδειγμα τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία, το Σεχέλ και τις χώρες του Περσικού κόλπου. Επιπλέον το 2017 το Προεδρείο ενέκρινε την διεύρυνση της λειτουργίας αυτού του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια από το 2018. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Πομιανόφσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να κάνω αυτή την παρουσίαση και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την ε, παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό που μας δίνει αυτή η ευκαιρία ετησίως. Μας δίνει τη δυνατότητα να κρατάμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο για τις δραστηριότητές μας. Και είναι και σημαντικό να ακούμε την υποστήριξη και να λαμβάνουμε υποστήριξη από τα, από τα μέλη για τις δραστηριότητές μας. Αυτή η σχέση μεταξύ του Ταμείου μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζεται και παγιώνεται μέσω του μηχανισμού διακυβέρνηση. Διότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Και έτσι υπάρχει μονίμως εκπροσώψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες μας. Και έτσι είναι ενημεροί για τις προτεραιότητές μας και λαμβάνουν τη λεπτομερή μας ε, εξαμηνία έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Το περασμένο έτος, το 2017, υπήρξε δυστυχώ ταραγμένο για τη δημοκρατία. Πολλές ε, κοινωνίες ε, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, ε, συγκρούσεις, σειράξεις, τοξικά αφηγήματα και απειλές για τη δημοκρατία. Απειλές για τη δημοκρατία που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ευρωπαϊκή γειτονία όπου παρέχουμε εμείς τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Ενώ οι προκλήσεις όλα ένα μεγαλώνουν, αποδεικνύεται διαρκώς πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη του Ταμείου μας και πόσο αξία προσφέρει η προσέγγιση μας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Ε, εγώ πρόκειται σύντομα να παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μας το 2017 με συγκεκριμένο τίτλο «Την υποστήριξη των ανθρώπων που παλεύουν για τη δημοκρατία» μπορείτε να λάβετε και εσείς αυτή την έκθεση και μπορείτε να τη βρείτε και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Όπως λέει ο τίτλος, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που μάχονται για τη δημοκρατία. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι οι άνθρωποι πράγματι βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών μας. Υποστηρίζουμε εκατοντάδες ανθρώπους και ομάδες. Πολλοί από αυτούς ε, διακινδυνεύουν τις ζωές τους ε, για να ε, προωθήσουν τις δημοκρατικές αξίες. Το 2017 ήταν άλλο ένα έτος μέσα στο οποίο παγιώσαμε τη θέση μας. Όπως είπαμε υπήρξαν ε, ήταν το τέταρτο έτος ε, επιχειρησιακή μας δραστηριότητας. Εμεί ξεκινήσαμε, υπενθυμίζω, το 2013, ενώ η απόφαση είχε ληφθεί το 2011. Κατά το διάστημα αυτό και κατά την παγίωση τη θέση μα ε, έχουμε καταστεί ένα σημαντικό οργανισμό για την υποστήριξη τη Δημοκρατία. Πέρυσι υποστηρίξαμε πάνω από 160 πρωτοβουλίε και ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας σε 20 χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς εστιαζόμασταν στην παροχή ε, χορηγιών στους πιο ενεργούς ε, ακτιβιστές ε, στην περιοχή, γύρω από την περιοχή μας αποδεικνύουμε πόσο σημαντική είναι η εντολή μας η προσθήκη αξία στη δημοκρατία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το Ταμείο δεν είναι το μόνο εργαλείο που υπάρχει στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων των κρατών μελών αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ένα ξεχωριστό μέσο για τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ μας, τη συμπλήρωση των κενών και το ότι θα μπορούμε να προσφέρουμε την επιπλέον υποστήριξη που αλλιώς δεν θα μπορούσε να παρασχεθεί. Στα τέλη του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενέκρινε την επέκταση των ε, επιχειρήσεών μας στα Δυτικά Βαλκάνια των δράσεών μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα υποστήριξη που θα καλύπτουν τρει βασικού τομεί: κοινωνία των πολιτών, ανεξάρτητα μέσα και πολιτικοί ακτιβιστέ και ειδικότερα νέοι. Όπω με την υπάρχουσα στήριξη, το Ταμείο μα θα εστιαστεί στην προσθήκη αξία και στην παροχή συμπληρωματική στήριξη σε άλλα προγράμματα υποστήριξη τη Δημοκρατία και φυσικά στήριξη η οποία θα επεκταθεί μέσω τη διαδικασία προσχώρηση στα Δυτικά Βαλκάνια στις ε, αντίστοιχε χώρες. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τρεις πρωτεύουσες, τέσσερις πρωτεύουσες στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό συνεχίζεται. Ήδη έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, και δραστηριές αποκρίσεις από τους μελλοντικού εταίρους μας. Η απόφαση ελήφθη μόλις το Δεκέμβριο πέρυσι. Πιο ευρέως για τις εργασίες μας ε, αισθανόμαστε ότι όλο και μεγαλύτερη σημασία αποκτά ο ακτιβισμός. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και το πώς εμείς υποστηρίζουμε τους ακτιβιστές μέσω του Ταμείου. Λαμβάνουμε λοιπόν πιο στοχευμένες αιτήσει και πολύ συγκεκριμένες ανάγκες που απαιτούν συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στις Βρυξέλλες ε, και στις πρωτεύουσες των χώρων, η οποία όλο ένα μεγαλώνει τόσο για το συμπληρωματικό μας ρόλο όσον αφορά την, τα προγράμματα υποστήριξης της δημοκρατίας, όσο και στην παροχή πολιτικής στήριξης προς εμάς για να εργαστούμε ε, πιο αποτελεσματικά. Οι χώρες ε, που είναι μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου και ο Καναδάς έχουν συμμετάσχει στον προπολογισμό μας. Η ετήσια χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας διασφαλίζει ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα και μας παρέχει επίσης ε, ε, θεσμική σταθερότητα. Ωστόσο, η συνεχής υποστήριξη στις προσπάθειές μας είναι κρίσιμη για να μπορέσουμε να έχουμε συνεχείς προσπάθειες και να συνεχιστούν η υποστήριξη μας προς τους ακτιβιστές. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι πολύτιμη η βοήθειά σας, ειδικότερα όταν είστε στις πρωτεύουσές σας και μπορείτε να εκφέρετε τις δικές σας γνώμες ε, στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στις ε, πρωτεύουσές σας. Η ετήσια έκθεση που έχετε μπροστά σας παρουσιάζει μια γενική εικόνα των διαφόρων πολιτικών περιβαλλόντων όπου λειτουργούμε από τα μεταβατικά μέχρι τα, και τα περιοριστικά μέχρι τα αυταρχικά καθεστώτα και τις ε, καταστάσεις σύραξης. Εξετάζει τις προκλήσεις που παρουσιάζει καθένα από αυτά τα περιβάλλοντα και δίνει παραδείγματα αποκρίσεων αποτελέσματα και μελέτες περιπτώσεων. Λόγω της διαφορετικότητας των περιοχών όπου εργαζόμαστε από τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοαφρική μέχρι την ανατολική εταιρική σχέση και πέραν αυτή, το Ταμείο υιοθετεί μια ευέλικτη και μη συμβατική προσέγγιση, προσαρμόζοντα την υποστήριξη στι διαφορετικέ συνθήκε. Επενδύουμε σε μεταρρυθμιστικέ ιδέε και στου ανθρώπου που τι στηρίζουν. Η ιδιαιτερότητά μα βασίζεται στην ικανότητά μα να λειτουργούμε σε δύσκολα, συχνά επικίνδυνα περιβάλλοντα, τα οποία δεν είναι προσπελάσιμα σε πολλούς χορηγούς. Μέσω της δικής μας στήριξης, αναφέρθηκε πριν από δύο μέρες ε, για την παροχή στήριξης, Είμαστε ένας ε, ταχύς μηχανισμός. Ε, ο μέσος χρόνος απόκρισης για επίγουσα στήριξη είναι δυο με τρεις εβδομάδες. Για τυπική κλασική βοήθεια 12 με 15 εβδομάδες από την αίτηση μέχρι την ε, παροχή της στήριξης. Μέσω τη στήριξή μα ε, αναπτύσσουμε τι ικανότητε των πολιτών και ενισχύουμε τι ανεξάρτητε φωνέ. Πολλέ από αυτέ τι φωνέ λένε τι δικέ του ιστορίε μέσω μια σειρά ε, προφίλ αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο που θα βρείτε μέσα στην έκθεση. Μέσω αυτή τη προσωπική διάσταση, σκοπό μα είναι να δείξουμε πραγματικά τον αγώνα και πώς έχουν πραγματικά οι συνθήκες στην πραγματική ζωή και πόσα πολλά μπορούν να επιτευχθούν με έναν απλό συνδυασμό μια μικρή στήριξη από ένα μικρό οργανισμό όπως το δικό μα και με την ισχυρή βούληση των ανθρώπων που βρίσκονται επί τόπου. Ενώ το περιβάλλον και η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με την περίπτωση, ε, παρατηρούμε ότι οι ισχυρέ δημοκρατίες είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασφάλιση της βιώσιμη ευημερία. Αυτοί οι ακτιβιστέ διακεντρέμουν τι ζωές τους για να αμφισβητήσουν κατασταλτικά καθεστώτα, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να προστατεύσουν την ελευθερία ομιλία ε, ε, και του συνεταιρίζεστε. Ε, και συχνά αντιμετωπίζουν εκστρατείε αμαύρωση που προσπαθούν να του εκφοβήσουν. Στην έκθεση θα βρείτε την ιστορία του Δημήτρου Μπουλάκ, ενό αιρετού αξιωματούχου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Χαρκίβ στην Ουκρανία και επικεφαλή ε, του Κέντρου Καταπολέμηση Διαφθορά ε, του Ταμείου μα, που αποκαλύπτει πρακτικέ διαφθορά και κατάχρηση δημοσίων οικονομικών στο Δήμο. Προφανώ δεν είναι αρεστό σε όλου. Το 2017 του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν ε, σωματικά πολύ άσχημα καθώς πήγαινε προς τη δουλειά του και δεν βρέθηκαν οι δράστες. περιπτώσει αν αυτές δείχνουν ότι οι ακτιβιστές, οι ακτιβιστές αυτοί διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε συνθήκες που διέπονται όχι από το κράτος δικαίου αλλά από τον νόμο του φόβου και της βιότητας. Στην Αίγυπτο έχουμε δει υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συλλαμβάνονται με ψευδείς ε, κατηγορίες ε, ότι υποτίθεται ανήκουν σε τρομοκρατικές μονάδες. Ε, σε τρομοκρατικέ ομάδε. Δεν θα το πιστεύετε, αλλά ένα δικηγόρο που ήρθε στο αστυνομικό τμήμα για να υπερασπίσει έναν ακτιβιστή επίση ε, συλλήφθηκε. Ο κατάλογο είναι τεράστιο, αλλά όλε αυτέ οι απειλέ, η παρενόχληση και η βία ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αποφεραίνουν αυτού του θαραλέου ανθρώπου. Σε χώρε όπω το Αζερβαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Αίγυπτο, η Ρωσία, όπου δεν υπάρχει χώρο για πολιτικό και ε, αστικό ακτιβισμό, το Ταμείο παρέχει στήριξη στις ομάδες υποστήριξης της δημοκρατίας ώστε να συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους παρά το δύσκολο νομικό και πολιτικό περιβάλλον. Στις ζώνες σειράξεων το Ταμείο μας ε, δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι πληθυσμοί που πλήττονται από τον πόλεμο και την αστάθεια δεν θα παραμεληθούν. Για παράδειγμα, στη Συρία το Ταμείο μα προσαρμόζει την υποστήριξή του σε ομάδε υπερασπιστή τη δημοκρατία και σε ακτιβιστέ για να καλύψουν τι ανάγκε του στο όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον. Τους βοηθάμε λοιπόν να παραμένουν δραστήριοι ώστε να μπορέσουν να παίξουν ρόλο στο μέλλον ε, εμπνέοντας ε, τον κόσμο με τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Παραλάμε το έργο της ε, στη χώρα, το Ταμείο μας υποστηρίζει διάφορες πρωτοβουλίες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές σε κοινότητες προσφύγων στο Λίβανο και όχι μόνο. Εγώ μόλις επέστρεψα την προηγούμενη εβδομάδα από το Λίβανο όπου συνάντησα διάφορους ε, ε, δικαιούχους ε, χορηγιών του Ταμείου μας που εργάζονται σε διάφορους τομείς σε ανεξάρτητες πλατφόρμες μέσων, οργανισμούς watchdog, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κτλ. Για παράδειγμα, επισκεφθήκαμε την πόλη της Τρίπολης στο Βόρα, όπου η μαζική άφηξη προσφύγων δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις και εκεί χρηματοδοτήσαμε έναν οργανισμό που ονομάζεται Lamsat World, που δημιουργεί μια κοινότητα η οποία παρέχει ένα μείγμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε νέους προσφύγους ώστε να μπορέσουν να χειραφετηθούν πολιτικά και πολιτιστικά με μακροχρόνιο στόχο να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί η ηγεσία μεταξύ των νέων, η αίσθηση της πολιτικής ηγεσίας ε, σε Συρίους πρόσφυγες όταν θα επιστρέψουν στη Συρία. Παρότι μας εμπνέει η δημιουργικότητα και η αφοσίωση όλων των εταίρων που έχουμε συναντήσει, μας ανησυχεί ε, το πόσο επιδονώνται οι νομικές και οικονομικές ε, ε, συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσουν οι ακτιβιστές της ΣΥΡΙ εκεί. Ένα σημαντικό τομέα όπου το Ταμείο μας παίζει σημαντικό ρόλο είναι η υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η έκθεση εξετάζει σε βάθος την υποστήριξη σε αυτά τα μέσα και στις δύο περιοχές και στις χώρες Ανατολικής Αντρικής σχέση στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Ο περιορισμό του τύπου παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. Περίπου το 1 τρίτο των πρωτοβουλειών υποστήριξη από το Ταμείο μα σχετίζονται με τα μέσα. Εμεί προσπαθούμε να αναπτύξουμε πόρου εκεί όπου μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη επίδραση και να καλύψουν κενά σε τομεί που δεν καλύπτουν άλλοι χορηγοί και η δική μας χρηματοδότηση βοηθά την ανάπτυξη των τοπικών μέσων ως ανεξάρτητων και αξιόπιστων και ποιοτικών ειδησιογραφικών πρακτορίων. Επίσης έχουμε επενδύσει σημαντικά σε καινοτόμες εργασίες για να συμβάλλουμε στην απόθεση της παραπληροφόρησης της Ρωσίας στις χώρες Ανατολικής Ιτρικής Σχέσης, ενισχύοντας τα ανεξάρτητα μέσα ρωσικής γλώσσας σε αυτές τις χώρες. Με περηφάνεια μου ανακοινώνω ότι πριν από δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε ένα νέο ταμείο, το Ταμείο Δημιουργικού Περιεχομένου, το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση σε ανεξάρτητα ε, ανεξάρτητου ιδιοσιογραφικούς ε, ρωσόφωνου οργανισμού στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και τώρα σιγά σιγά γίνεται ένα σημαντικό ανεξάρτητο ε, μέσο που χρηματοδοτείται από πολλού χορηγού με σκοπό να υπάρχει πολυφωνία και ισορροπία στο χώρο των ανεξάρτητων ιδιοσιογραφικών μέσων ρωσική γλώσσα. Όλα ξεκίνησαν με μια έκθεση του 2015 του Ταμείου που συνιστούσε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα για την απόθεση των προσπαθειών προπαγάνδας της Ρωσίας στην περιοχή. Για να συνοψίσω, είναι δύσκολε εποχέ για τη δημοκρατία. Οι απειλέ και οι προκλήσει είναι μεγαλύτερε από ποτέ μετά τα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Κρεμλίνο πραγματοποιεί πληροφοριακό πόλεμο μέσω ε, διαρροών παραπληροφόρηση, προσπαθώντα να εκθέσει τι ελλείψει των δυτικών δημοκρατιών, ε, προωθώντα ένα αφήγημα ότι οι δυτικέ δημοκρατίε είναι το ίδιο διαφθαρμένε όσο και το ίδιο κατασταλτικό ε, προπαγανδιστικό καθεστώς της Ρωσίας. Δεν υπάρχουν γρήγοροι τρόποι διόρθωσης ή μεταρρύθμισης. Δεν θα γίνουν μέσα σε μια νύχτα. Αλλά κάτω από την επιφάνεια η στήριξη του Ταμείου μας συμβάλλει σημαντικά στο να αλλάξει το τοπίο. Στην καθημερινή μας δουλειά στο Ταμείο μας ε, έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με ακτιβιστές που αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολο είναι να ζει σε μια δημοκρατία και οι οποίοι επιθυμούν να μαχηθούν και να θυσιαστούν για να αλλάξουν τις κοινωνίες τους και να γίνουν πιο δημοκρατικές. Και εμείς παραμένουμε μετακίνητοι στην πεποίθησή μας ότι έχουμε ηθικό καθήκον να δείξουμε ε, αλληλεγγύη στους ανθρώπους που μάχονται για τη δημοκρατία, για τα ιδανικά της. Ελπίζω ότι ε, θα διαβάσετε με μεγάλη απόλαυση τις ιστορίες ε, αλλαγής και θάρρος που θα υπάρχουν στην εκθέσή μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση σας για να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Γκζίπ πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δευθυντά, σας ευχαριστώ ειλικρινά για την παρουσίασή σας και για την περιγραφή αυτή στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Ταυτόχρονα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουν περάσει μόλις πέντε χρόνια από την ίδρυση του Ταμείου και μία επτά ετία από την αρχική πρόταση για τη δημιουργία του Ταμείου. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο λοιπόν για τη Δημοκρατία έχει αρχίσει να λειτουργεί και ε, έχει περάσει σε μία ε, ταχύτητα μεγαλύτερη. 33 χώρες, είπατε, ε, συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο μαζί και ο Καναδάς. Και είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές δηλαδή οι χώρες που συμμετέχουν. Ε, στη συνέχεια καταφέραμε ε, να επιτύχουμε ε, μια ισορροπία στις διάφορες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούμε και προς Ανατολάς αλλά και προς το Νότο ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν η ισορροπία στην εργασία του Ταμείου και πολύ διαφορετικές οι προκλήσεις βέβαια στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία είναι πάρα πολύ ταχύ στην αντίδρασή του στις διάφορες εξελίξεις και στα γεγονότα που παρατηρούνται. Σε αντίθεση με τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρειάζονται μάλλον περισσότερο χρόνο για να αντιδράσουν και για να έχουν αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία υποστηρίζει και βοηθάει την κοινωνία των πολιτών επί τόπου. Και αυτό είναι τους λόγους για την καλή φήμη του Ταμείου. Είναι πραγματική επιτυχία, ε, ακτινοβολεί το Ταμείο και σας ε, συγχαίρω γι' αυτό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία είδε την εντολή του πέρυσι να επεκτείνεται έτσι ώστε να καλύπτει και τα Δυτικά Βαλκάνια, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό από τη σκοπιά ε, της διαδικασία σύνδεσης και προεταξιακή διαδικασία που διανύουν τα κράτη αυτά. Είναι πολλές οι χώρες που ενδιαφέρονται, που υποφελούνται και θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο κόσμος προβληματίζεται στις χώρες αυτές ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι πάντα εύκολο οι ερωτήσεις αυτές να βρίσκουν απάντηση για των ε, επίσημων διάβλων. Οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε το δικό σας ταμείο και σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά πράγματα. Ε, για τα οικονομικά του Ταμείου. Πώς έχουν εκεί τα πράγματα. Και πώς έχει η απόσπαση των εμπειρογνωμόνων ε, από τα διάφορα κράτη-μέλη στα δικαιούχα κράτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στρεβίτσιος. Α, συγγνώμη. Προηγουμένως η κυρία Φωτίγκα ζητώ συγγνώμη. No problem, Petra. <laughs> Ναι, δεν πειράζει. Δεν έχω πρόβλημα να είμαι πρώτη, δεύτερη, κανένα πρόβλημα. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή σας ε, την ε, παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης. Ως ήθιστε ενώπιον της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Και ενώ εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω εδώ στην καθημερινή μου δραστηριότητα εδώ στο Κοινοβούλιο ότι όντως ε, επωφελούμε από την εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία για την ε, βοήθεια για την οποία θέλω να σας ευχαριστήσω σας και τους συνεργάτες σας για τη μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε. και να προετοιμάζουμε καλύτερα τις εκθέσεις μας καθώς και τις στρατηγικές μας, τα στρατηγικά μας ανακοινοθέντα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ το Ταμείο για την ταχύτητα τα προσαρμοζόμενη ε, εργασία σας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έχετε εστιαστεί, όπως μας είπατε, και στα Δυτικά Βαλκάνια, κάτι το οποίο είναι αναποφευκτό και το στηρίζουμε όλοι μας. Αλλά έχετε και την δυνατότητα να παρατηρείτε τις αλλαγές και να βρίσκεται νέους τρόπους και μεθόδους λειτουργίας. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα για αυτή την πλατφόρμα όπου ε, μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο από διάφορα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και πιστεύω πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος Η ερώτησή μου αφορά την οικονομική σταθερότητα μετά από το Brexit. Ε, ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την κατάσταση. Ξέρω περίπου ποια είναι η κατάσταση, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω εάν υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω εξελίξεις, ενδεχόμενες εξελίξεις. Καθώς Επίσης, ε, αν υπάρχει ενδιαφέρον για ε, επέκταση σε ρωσόφωνα μέσα και επίσης κατά πόσο είναι ωφέλιμη μια τέτοια δραστηριότητα. Ευχαριστώ τώρα κύριο Σωστρεβίτσιο, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει και που μίλησα αργότερα δεν πειράζει. Θέλω να συγχαρώ τον Γιάννη Πολιανόφσκι και να συγχαρώ και το Έλμαρ Μπροκ. Ναι, Έλμαρ, για σένα λέω. αναγνωρίζετε το έργο σου στο σωστό τόπο και χρόνο. Γιατί ήταν από τους εμπνευστέ ε, αυτής της σημαντικής ε, διοργάνωσης, αυτού του σημαντικού θεσμού του Ταμείου. Κοιτάξτε, ζήτηση υπάρχει στην αγορά. Υπάρχουν χώρες δηλαδή ε, όπου δραστηριοποιείστε και καλύπτεται που δεν διακρίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθεροτυπία, την ελεύθερη διακυβέρνηση κτλ. Υπάρχει χώρος δηλαδή για να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο, να το ανεβάσουμε αυτό των κρατών και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δώσουμε μία όθηση για διάφορες διεργασίες που χρειάζονται πολλές φορές διαφόρων ειδών. Εσείς έχετε μια θέση πλεονεκτική. Γιατί αντιδράτε γρήγορα, είσαστε ευέλικτοι και πολύ εστιασμένοι στην πρακτική προσέγγιση όταν θέλετε να υποστηρίξετε τη συνεργασία σε πολλούς φορείς και πολλές δομές. Ακτιβιστές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμοί περιμένουν από σας συνεχίστε ε, με αυτό το μοντέλο και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα, είμαι βέβαιος. Χαίρομαι πάρα πολύ και εκτιμώ το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε να ε, διηγούνται την προσωπική τους ιστορία οι, ε, οι, ακτιβιστές. Συγγνώμη. Έχουν αυτό το αφήγημα το οποίο ε, πολύ εκτιμούμε με προσωπικές ιστορίες και πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι μελλοντικοί ε, βραβευθέντες ε, του βραβείου Ζαχάροφ. Είναι ποιοτικό το αποτέλεσμα, ήδη φαίνεται από τις πρώτες προσπάθειες. Όπως είπατε, έχετε επεκτείνει τις δραστηριότητε σας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, πράγμα που χρειάζεται και καλή σας τύχη εκεί, και στην Τουρκία. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για την Τουρκία. Γιατί σε τούτη εδώ την Επιτροπή αφιερώνουμε πολύ χρόνο ε, στη συζήτηση για διάφορες πτυχές της κατάστασης στην Τουρκία. Και θα ήμουν πραγματικά περίεργος και θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι κάνετε στην Τουρκία. Έχετε σχέδια να ξεπεράσετε την οροφή των 20 κρατών στα οποία δραστηριοποιήσετε σήμερα. Και καλή τύχη για τις επόμενες προσπάθειες σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσεριτς. Thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξοχότατε, κύριε Πρέσβη Πομιανόφσκη, θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Ας αρχίσω από μια προφανή δήλωση, αλλά εσείς και το ταμείο σας πραγματικά δεν είστε καθόλου περιττή. Βλέπουμε πόσο περιορίζεται ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στα διάφορα κράτη. Είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί ε, μια τέτοια οργάνωση σαν τη δική σας για πολύ καιρό ακόμα. Που βασικά αυτό είναι δυσάρεστα νέα. Τα ευχάριστα είναι ότι ό,τι δουλειά κάνετε είναι εξαιρετική. Όλο αυτό το εγχείρημα με αυτόν τον τρόπο, με την ευελιξία, με την ταχύτητα στην αντίδραση ε, και με μικρού επίπεδου χαμηλή χρηματοδότηση μέσα είναι πολύ σημαντική. Ε, εξίσου σημαντική με τη μακροοικονομική βοήθεια και ε, τα λοιπά που χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Χαιρόμαστε φυσικά για την επέκταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Πραγματικά υπήρχε ευρεία εδώ συνένεση στο Κοινοβούλιο ότι κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο και έπρεπε να γίνει. Αλλά αυτό που θα πρέπει τώρα να εξασφαλίσουμε είναι να υπάρχουν οι σωστοί απαραίτητοι πόροι για να μπορεί το Ταμείο να ανταποκρίνεται στην αποστολή του. Και έχω τώρα κάτι που είναι μισή ερώτηση, μισή παρατήρηση. Λυπούμεθα πάρα πολύ που υπάρχουν σημαντικά κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν δώσει τις συνεισφορές τους ακόμα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Και επίσης λυπάμαι για το γεγονός ότι απουσιάζουν οι συνάδελφοι από τις χώρες αυτές, οι οποίες είναι Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία. Και θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας διαφωτίσουν οι συνάδελφοι αν ήταν πάροντες γιατί δεν δίνουν τα λεφτά ε, τα κράτη. Αν θέλουμε να έχουμε κάποια ισορροπία μεταξύ Νότου και ανατολή στην Ευρώπη, Χρειαζόμαστε πόρους από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν περισσότερο και ενδιαφέρονται περισσότερο για τους τομείς αυτούς. Αν έχετε ελαφρυντικά στοιχεία που να δικαιολογούν γιατί το κάνουν αυτά τα κράτη, να μας το πείτε. Αλλιώς θα ήθελα να ακούσω Επίσης, εμείς ως ομάδα, οι πράσινοι, ενδιαφερόμαστε πολύ ε, για την επέκταση της δραστηριότητάς σας ε, υπέρ της και υπέρ της πάταξης της διαφθοράς. Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα. Εκεί μπορεί να γίνει διαφορά, ιδιαίτερα σε καταπιεστικά καθεστώτα. Το 1 τρίτο των μικρών ε, επιδοτήσεων πηγαίνουν σε χώρες που έχουν τέτοιου είδους κατασταλτικά καθεστώτα. Θέλω να σας εθαρρύνω να αναπτυχθείτε ε, προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πιάνουν τόπο τα χρήματα και ε, στις κοινωνίες και μπορεί να μας δώσει και κάποια δυνατότητα εισόδου εκεί για να έχουμε μια κοινωνία των πολιτών πιο πολιτικοποιημένη σε αυτούς τους τομείς. Τα υπόλοιπα μπορούμε όλα να τα συζητήσουμε διμερώς ξεχωριστά Πάντως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είστε εδώ και ότι υπάρχει αυτός ο οργανισμός και έχει αυτό το έργο. Ευχαριστώ κύριος Βέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον uh, κύριο Πρέσβη για την εργασία του, για τον εκδημοκρατισμό της των, των ανατολικών και νοτιών γειτόνων μας. μπορούμε να έχουμε επαφή με άτυπες ομάδες που δεν θα ήταν επιλέξιμες ε, ε, για χρηματοδότηση από τα προγράμματα της Ένωσης. Φαντάζομαι πως ήταν δύσκολο πολλές οι προκλήσεις για τη δημοκρατία και πως είπατε το 2018 θα είναι δύσκολο και αυτό. Και ελπίζω ότι με τους ε, διάφορους εταίρους ε, θα συνεργαστούμε για να ε, ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με την βιωσιμότητα και την ε, ιδιοποίηση των project που, που, που στηρίζει το Ταμείο. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της δημοκρατίας. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για πρωτοβουλίες που αφού χρηματοδοτήθηκαν μπόρεσαν να γίνουν βιώσιμες, να σταθούν μόνες τους ή, με πάση περιπτώσει, να μειώσουν την εξάρτησή τους από εξωτερική βοήθεια. Μάλιστα τώρα η κυρία Χάρμς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και από τη δική μου πλευρά να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα στις δραστηριότητες ε, του Ταμείου για τη Δημοκρατία. Νομίζω πως είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που λάβαμε να το φτιάξουμε χάρη στον κύριο Μπούζεκ και όσους ε, στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία αυτής της συνεδρίασης για να συζητήσουμε για ένα θέμα με το οποίο εγώ διαρκώς εργάζομαι. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω είναι Πώς σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναχαιτήσει την ρωσική προπαγάνδα και όλες τις σχετικές εξελίξεις. Έχουμε συμφωνήσει με αυτήν την έκθεση της ε, κυρίας Φωτίγκα πριν από λίγο καιρό ότι η εγκαθίδρυση ανεξαρτήτων μέσων και η διευκόλυνση ποιοτική ανεξάρτητης δημοσιογραφίας είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες που θα έπρεπε να στηριχθούν. Εγώ διαπιστώνω ότι ιδιαίτερα στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες εταίρους οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι δεν ε, αντιμετωπίζουν μόνο πολιτική πίεση, αλλά και την ε, αδυναμία επιβίωσης με βάση τη δουλειά τους, πράγμα το οποίο κανονικά εμείς πολύ το εκτιμούμε όταν τους ε, συναντούμε. Οπότε... Ε, κανονικά θα έπρεπε να μπορούν να είναι βιώσιμοι μετά από σύντομη στήριξη, χρονική στήριξη ε, από την Ένωση από άλλους. Όμως, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι και πολύ πιθανό να μπορούν να σταθούν μόνοι τους αυτού του είδους οι δημοσιογράφοι. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα. Γιατί, από όσο εγώ γνωρίζω, και καλύτερη μου συμβουλή θα ήταν να στηρίξουμε ποιοτική δημοσιογραφία σωστή ενημέρωση και ανεξάρτητα μέσα και ανεξάρτητους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε αυτό το γύρο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις θα κάνω, μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουμε ότι αυτός ο θεσμός υπάρχει εδώ και λίγα χρόνια και ακόμα είναι στη φάση της δημιουργίας του. Θέλω να πω όμως και στους υπαλλήλους ότι πραγματικά το έχετε φέρει σε πέρας εξαιρετικά δεδομένων των δυσκολιών των γνωστών που είχατε. Και γι' αυτό χαίρομαι για αυτά που ακούω. Ήταν δική μας ιδέα πράγματι να γίνει κάτι έτσι ώστε εκεί που είναι δύσκολο επίσημα να υπάρχει μια δράση. Να βοηθήσουμε. Να διευκολύνουμε περισσότερα τα πράγματα εκεί που δυσκολεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επίσημη χρηματοδότηση και την τυπική. Και ουσιαστικά είναι ε, ουσιαστική βοήθεια και ουσιαστική βοήθεια ε, στην κοινωνία των πολιτών, συγκεκριμένη ε, ε, βοήθεια σε επίπεδο πολιτών και όχι διαπληκτισμοί με την ηγεσία και συγκρούσεις, που θα ήταν λάθος. Σε χώρες που δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ή πολύ λίγη δημοκρατία και κράτος δικαίου. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τώρα, πάμε στα Βαλκάνια, ή πού πάμε στα Βαλκάνια, να μην το θεωρήσουμε ρουτίνα. Ένα να κάνουμε αυτή τη δύσκολη δουλειά και σε καθεστώτα που μπορεί να είναι δικτατορικά. Με όλες τις απειλές και τις προκλήσεις. Σωστό είναι αυτό που είπε ο κύριος Μέσεριτς προηγουμένως. Ε, σχετικά με την ισορροπία. Μέχρι τώρα καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Και ο κύριος Μέσεριτς είπε κάτι σημαντικό. Το ταμείο αυτό ζει από την ετήσια χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και άλλων κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κάθε χρόνο χρειάζεται αυτή η υποστήριξη και δυστυχώς οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, συμμετέχουν ελάχιστα έως καθόλου μέχρι στιγμής ε, στη χρηματοδότηση, παρόλο που είναι μέλη του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Όλα τα κράτη-μέλη είναι μέλη στο Ταμείο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά η συμμετοχή στη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ ετεροβαρής. Και μήπως μπορούν να μας βοηθήσουν οι συνάδελφοι για να χτυπήσουν κάποιες πόρτες στις πατρίδες τους και να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις τους να δράσουν γιατί αν δούμε τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, καλό θα ήταν και χρήσιμο να υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή των νοτίων κρατών, δεδομένων των αναγκών και των συνθήκων που επικρατούν εκεί. Οπότε καλό θα ήταν να το ξανασκεφτούμε και εμείς, Πρόεδρε, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για να συνεννοηθούμε περισσότερο με τις χώρες του Νότου για να κάνουμε κάτι υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην άμεση γειτονία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε Πομιανόφσκι, παρακαλώ, για να απαντήσετε. Thank you, Chair. Thank you Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους ε, όσους συμμετείχατε σε αυτή την ε, συζήτηση. Καταρχάς, Ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ακούσαμε τόσα καλά λόγια και τόση εκτίμηση για την εργασία μας. Είναι υπέροχο να έχουμε την υποστήριξή σας. Οι ερωτήσεις σας είναι ιδιαίτερα κέρυες όλες και βέβαια είναι και κομμάτι των καθημερινών μας προβληματισμών. καλύτερη μεθοδολογία μου φαίνεται είναι να απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν οι ερωτήσεις. Να απαντήσω στον κύριο Ξύμπ για την ε, ε, συλλογή κονδυλίων και την γενικότερη στήριξη από τα κράτη-μέλη. Καταρχάς, όντω είναι αλήθεια ότι η παροχή για τον ε, χρημάτων για τον προπολογισμό του Ταμείου δεν είναι η μόνη βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε από τα κράτη-μέλη. Ε, από τη Δανία, ας πούμε, λάβαμε μια υποστήριξη με, έναν, με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που μας βοήθησε ε, με μία απόσπαση δηλαδή ενό Ε, Επίσης, ε, λαμβάνουμε σημαντική βοήθεια από τις πρεσβείες ε, των κρατών μελών στις χώρες όπου μεταβαίνουμε και έχουμε τις δικές μας επαφές ή κάνουμε τις αποστολές μας το πρώτο σημείο επαφής λοιπόν είναι πάντα η αντιπροσωπεία της Ένωσης. Μας δίνουν μεγάλη υποστήριξη, αλλά επίση τα κράτη-μέλη. Το κρατών ε, Πολωνία, Γερμανία, Κατοχώρε, ε, Σουηδία, Νορβηγία και άλλοι, για να μην του αναφέρω τώρα όλου, αλλά πολλοί αντιδρούν αμέσως στα αιτήματά μας είτε για ενημέρωση είτε και για άμεση υποστήριξη υπό τη μορφή διοργάνωση συνεδρίων, επαφών, οργάνωση ε, των μεταφορών και πολλούς και διάφορους τρόπους. Αυτό το είδους η στήριξη και αναγνώριση είναι εξαιρετικά σημαντική και το νιώθουμε και τόπου. επίσης στις πρεσβείες στρεφόμαστε οποτεδήποτε υπάρχει κάποια πρόκληση ασφάλεια. ε, ή όταν ε, κινδυνεύουν ας πούμε οι ε, άνθρωποι με τους οποίους είμαστε σε επαφή ή που έχουν λάβει υποστήριξη από εμά, τονίζουμε και σηματοδοτούμε τις πιέσεις και τις απειλές που μπορεί να δεχτούν οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτή η βοήθεια είναι πολύ σημαντική. Τώρα όπως οποιοδήποτε άλλος οργανισμός ε, μπορούμε πάντοτε να θέλουμε και άλλα και όσον αφορά το συγκεκριμένο ταμείο όπως αναφέρε ο κ. Μπρόκ, ο πρόεδρός μας αλλά και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτές έχουμε να αντιμετωπίσουμε έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη Δηλαδή αυτά των οποίων η γεωγραφική τοποθεσία είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και δίνουν περισσότερο από τα νότια κράτη. Ως προς αυτό, οποιαδήποτε υποστήριξη μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων, μέσω άμεσων επαφών με τους υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων, των σχετικών αποφάσεων, Οποιαδήποτε λοιπόν βοήθεια και υποστήριξη μπορεί να υπάρξει είναι ευπρόσδεκτη γιατί χρειάζονται συνέχεια περισσότερα χρήματα. Τα περισσότερα κονδύλια αποτελούν την εγγύηση ότι μακροπρόθεσμα θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ευέλικτη βοήθεια και να σχεδιάσουμε τι στρατηγικέ μα για μακρύτερε χρονικέ περιόδου από ότι ένα-δύο χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μελλοντική επιτυχία του Ταμείου. Μετά το Brexit σταθερότητα του ταμείου μας. Για την ώρα δεν απειλείται το ταμείο. Έχουμε λάβει πολύ θετικά μηνύματα από αυτούς που αναλύουν ε, την κατάσταση, ε, ιδιαίτερα την, ε, Ευρωπαϊ... την... το κονδύλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ταμείο μας Φαίνεται ότι υπάρχει υποστήριξη από εσά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι αυτό θα προστατέψει τον λειτουργικό προπολογισμό του Ταμείου μα από οποιασδήποτε δυσκολίε στο μέλλον. Όσον αφορά τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου συγκεκριμένα, η ερώτηση αυτή τέθησε σε μια από τι συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη σημαντικό ε, ε, συνεισφέρον στον προπολογισμό του Ταμείου μα. Ε, πολλά εκατομμύρια έχει καταβάλει και ρωτήθηκε τι θα γίνει ε, μετά το Brexit. Η απάντηση ήταν σαφής ότι το ε, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το Ταμείο για την Δημοκρατία είναι Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Δημοκρατία και όχι ε, Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία. Γι' αυτό και ε, είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι θα συνεχίσει η Βρετανική κυβέρνηση να υποστηρίζει το Ταμείο μας. Μάλιστα, η Βρετανική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην παροχή κονδυλίων για να στηριχθούν τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και να απόθυθει η ρωσική προπαγάνδα, να αναχαιτιστεί στην ανατολική εταιρική σχέση, αλλά και αλλού. Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ετησίω. Τώρα, για την κυρία Φωτίγα και για τα ρωσόφωνα μέσα. Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε άμεσα αποτελέσματα που συμβαίνουν εν μία νυχτή, αν και ήδη δουλεύουμε εδώ και δύο χρόνια στο τομέα αυτό. Είναι πολύ σκληρή δουλειά και πρέπει να δεχτούμε όλοι μας ότι έχουμε ξεπεράσει ορισμένε ε, περιπτώσεις όπου οι ειδικοί στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο τομέα ε, είχαμε ε, εκπροσώπους στη Μόσχα όπου ε, η κυρία Μάριν μας έδωσε εξαιρετικά ε, περιστατωμένη ανάλυση για το πόσο Πούτιν θεωρεί να, θέλει να επεκτείνει την επιρροή του στις γειτονικέ χώρες αλλά και στην ίδια του τη χώρα και αυτό το παραβλέψαμε τότε. Ε, ε, σήμερα θα είχα αντιδράσει τελείως διαφορετικά, αλλά το 2010 δεν το κάναμε αυτό. Για να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτή την καθυστέρηση, και όλες αυτές τις ε, διαδικασίες που έγιναν χρειάζεται σταθερή και μακρόπνοη δέσμευση για δράση. Τα σημαντικά και καλά νέα είναι ότι έχουμε ιδέες, έχουμε δημιουργικό κόσμο που δουλεύει διαρκώς, ε, προβληματίζεται, σκέφτεται ε, και έχουμε ήδη σημαντικές επιτυχίες. Τρεις πρωτοβουλίες που συστήθηκαν από την έκθεση του Ταμείου μας το 2015 ως προς αυτό για την ε, δημιουργία ενός κόμβου ανταλλαγής ρωσόφωνων νέων. Έχει έδρα στην Πράγα και έχει διάφορες εξόδους που συνδέονται με αυτό το κόμβο. Δουλεύει, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Έχουμε μια για δημιουργικές παραγωγές που δεν είναι άμεσα πολιτικού χαρακτήρα, αλλά που είναι ανεξάρτητες ε, διέξοδοι για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του ακροτηρίου με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα έκαναν με έναν περιορισμένο προϋπολογισμό. Δεν μπορούν ας πούμε, να φτιάξουν ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ ή ε, σοου ε, ή προγράμματα παιδικά που θα ήθελαν να το κάνουν, έχουν εξαιρετικές ιδέες, αλλά ο προπολογισμό δεν το επέτρεπε. Οπότε Εκεί έχουμε ένα τα κονδύλι για περιεχόμενο που στηρίζει τέτοιου είδου παραγωγέ, ήδη λειτουργεί και τα αρχικά αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα. Οι ε, συμμετέχοντες διαπιστώνουν ότι αυξάνεται και το ακροατήριό τους και η θεματικότητά τους και αυτή είναι πολύ θετική τάση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριος Τρεβίσιος που είπε ότι δεν υπάρχει έλλειψη ζήτησης. Πράγματι, το βλέπουμε αυτό καθημερινά, ότι παίρνουμε πάνω από χίλιες αιτήσει ε, ε, ετησίως. Τις διαβάζουμε όλες πολύ προσεκτικά, έχουμε επαφή με τους διάφορους φορείς και χρηματοδοτούμε σχεδόν το 10% όλων αυτών. Είναι δύσκολο λοιπόν όταν πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε τόσες πολλές ε, σπουδές αιτήσει και ανάγκες. Και όσον αφορά την ιδιοποίηση, την οικειοποίηση του, των προγραμμάτων αυτών, θα πρέπει να πω ότι το λειτουργικό επιχειρησιακό μοντέλο που βασίζεται απλά στη ζήτηση, στις τοπικές πρωτοβουλίες που γίνονται ούτως ή άλλως, άσχετα από το αν θα πάρουν τη δική μας στήριξη ή όχι, αυτοί οι άνθρωποι είναι δραστήριοι. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ότι το θέμα της τοπικής ιδιοποίησης των ε, πρωτοβουλειών είναι ε, αυταπάντητο και ότι ούτως ή άλλως χρηματοδοτούμε, όπως σας είπα, πρωτοβουλίες που θα γίνονταν ούτως ή άλλως. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις. Το Ταμείο, επειδή έχει μικρό προπολογισμό, δημιουργήθηκε ως ένας συμπληρωματικός μηχανισμός για να καλύψει τα κενά. Σημαίνει αυτό ότι η στήριξη η δική μας σπανίως ή σε πολύ λίγες περιπτώσεις επαναλαμβάνεται. Συνήθως στοχεύουμε στο να δώσουμε εμπειρογνωμοσύνη αλλά και συγκεκριμένη γνώση και δυνατότητες στους δικαιούχους μας, ώστε να ζητήσουν πιο μακροπρόθεσμη στήριξη αλλού, από πιο παραδοσιακούς δωρητές. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο και να δώσουμε γρήγορη και μη συμβατική στήριξη. Όμως όταν έχει πια ε, στηριχτεί, στηθεί το project, μπορεί να ζητήσει και Πολλοί μάλιστα έχουν ζητήσει ε, και με επιτυχία ε, χρηματοδότηση από την Ένωση, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από τις κατοχώρες και συνεχίζουν με επιτυχία τη δουλειά τους με πιο σταθερά και πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα και στο σύστημά μας ε, παρακολούθησης καταγράφουμε κάθε τέτοια επιτυχή πρωτοβουλία. Σε σχέση με το θέμα της Τουρκίας, έχουμε και εκεί project, αλλά για προφανείς λόγους δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί το περιβάλλον δεν είναι καθόλου εύκολο. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν τα βλέπετε στο site μας. 30% περίπου από τα project μας δεν φαίνονται στο site μας. Όταν διαβάζετε λοιπόν την έκθεση και όταν διαβάζετε το website, να θυμάστε ότι το 30% των project δεν αναφέρονται για πολύ σημαντικούς λόγους. Για την ερώτηση που αφορούσε τους σπόρους για τον Νότο. Ανέφερα ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στο γεωγραφικό βόρα και το γεωγραφικό νότο της Ένωσης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερη ισορροπία. Ακούμε κάποιες εξηγήσεις ότι η προσφυγική κρίση έχει τόσο πολύ ε, ταράξει τις χώρες αυτές που δεν έχουν χρήματα να προσφέρουν. Η μόνη χώρα που είναι ακόμα μπορεί και συμβάλλει είναι η Ισπανία, από αυτές που βρίσκονται στον Νότο. Και πρόσφατα είχαμε και μια μικρή συμβολή από την Κύπρο. Υπάρχουν μια, κάποια πρώτα σημάδια δηλαδή ότι τα καταφέρουν, αλλά χρειάζονται περισσότερα να γίνουν ώστε να είναι πιο ισορροπημένη η συμβουλή στον προπολογισμό του Ταμείου. Ήδη απάντησα στον κύριο Βέντα και στην ερώτησή του για την ε, ε, ιδιοποίηση των project και την κυρία Χάρμας να πω ότι έχετε δίκιο. Εμείς θεωρούμε ότι η αναχέτηση της προπαγάνδας με άλλη προπαγάνδα δεν είναι τρόπος ε, λειτουργίας. Γι' αυτό ο τρόπος να, να, μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τα τοξικά μέσα του Κρεμλίνου είναι να εγκαθιδρύσουμε από ε, πλουραλιστικά μέσα. Αυτό που είναι εναντίον μας δεν είναι μόνο η προπαγάνδα του Κρεμλίνου, αλλά είναι και η τοπική κατάσταση. Για παράδειγμα, η κατοχή των μέσων, ας πούμε, στην Ουκρανία από ολιγάρχες. Η αγορά των μέσων δεν λειτουργεί ε, ε, γι' αυτό και η μακροπρόθεσμη υποστήριξη από πλευρά τη Ένωση στα ανεξάρτητα μέσα είναι κρίσιμη, γιατί μετά μόνο με βραχυπρόθεσμη στήριξη δεν μπορούμε να ε, βασιζόμαστε στι τοπικέ ε, δυνάμει. Δεν είναι μια πορεία που θα διαρκέσει δύο-τρία χρόνια. Χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα 10-15 ετών για να στηριχθούν τα ανεξάρτητα μέσα. Το ίδιο βλέπουμε και στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να προστατευθούν και να παγιωθεί η ελευθερία τύπου και έκφραση στις χώρες αυτές, η ελευθερία των μέσων. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, πολλά, πολύ περισσότερα από τη δική μας δουλειά του Ταμείου. Συνεχιζόμενη στήριξη λοιπόν από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι απαραίτητη. Και τέλος, σε ευχαριστώ Έλμαρ Ευχαριστώ τον πρόεδρό μας που είπε λίγα λόγια συγχαίροντάς μας με αυτή την ευκαιρία της πέμπτης ε, επαιτίου από την ίδρυση. Ε, προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε λειτουργικοί χάρη στη δική σας σοφή Προεδρία και χάρη στην ιδιαίτερα πρικισμένη ομάδα που έχει το Ταμείο μας. Όμως η ανέβρεση κονδυλίων είναι ζήτημα για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μακροπρόθεσμα την σταθερότητα. Γι' αυτό είναι και το τελευταίο μου σχόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουμιανόφσκη. Για να κλείσουμε, έχω τη χαρά να σας πω ότι ε, η ομάδα ενίσχυσης δημοκρατίας στις 27 Ιουνίου διοργανώνει εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εορτάσει ε, την πέμπτη επέτειο από την ίδρυση του Ταμείου. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα, ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου. Dear uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας και παρακαλώ τους προσκεκλημένους που αποχωρούν να το πράξουν ησύχως. Ακολουθεί λοιπόν στη μερίσια διάταξή μας ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ζόραν Πάζιν, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό δικαιοσύνης του Μαυροβουνίου. Καλωσορίσατε θερμά ε, στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα επίση να καλωσορίσω τον πρέσβη, κύριο Μπόγιαν Σάρκιτς και την κυρία Βέσνα Μέντενιτσα, πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μαυροβουνίου. Υπουργέ Πάζιν, τα Δυτικά Βαλκάνια και το Μαυροβούνιο ιδιαίτερα προχωρούν προς την πλήρη ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχετε φτάσει στον πρώτο στρατηγικό σας στόχο, ε, εντασσόμενοι πέρσι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στρατηγική ε, για τα Βαλκάνια και ε, διάσκεψη στη Σόφια, τα μάτια στραμμένα όλων στο 2025. Η χώρα σας ε, πρωτοπορεί σε αυτό το μαραθώνιο. Ε, μαραθώνιος που δεν έχει τόσο χρονικά κριτήρια, αλλά επίδοση ως κριτήριο. Και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς νομικιστική, αλλά και ε, δηλώνει ότι στενίζεστε αξίες και αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν να σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει αποστολή αντιπροσωπεία στο Μαυροβούνιο για την παρατήρηση των προεδρικών εκλογών στις 15 Απριλίου. Η αποστολή αυτή θα έχει επικεφαλή στον συνάδελφο κύριο Καστάλντο Λοιπόν, κύριε Πάζιν, σας δίνω το λόγο για να μας πείτε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την ε, ένταξη της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κριστέα, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εκ μέρου τη κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και προσωπικά που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθύνω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια εξαιρετική περίσταση για μένα και καλή ευκαιρία για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του Μαυροβουνίου και να κάνω μαζί σας μια ανοιχτή συζήτηση που θα οδηγήσει σε συμπεράσματα τέτοια που θα βοηθήσουν ε, την πορεία της χώρας μου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής του Μαυροβουνίου είναι σαφείς. Ε, μέλος στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλές σχέσεις γειτονίας. Μέχρι στιγμής έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις ε, που υπάρχουν ε, καθοδόν για την υποστήριξη αυτών των στόχων. Να υπενθυμίσω ότι το να γίνουμε μέλη στο ΝΑΤΟ δεν ήταν κάτι απλό. Υπήρξαν κάποια εμπόδια. Ωστόσο, με τι δικέ μα δυνατότητε και με την στήριξη των δικών μα εταίρων, καταφέραμε να υπερβούμε, να υπερπηδήσουμε τι αντιστάσει που υπήρξαν και που έτειναν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα μα. Μια από αυτέ εμφανίστηκε την, ημερία, την ημερομηνία των δικών μα εκλογών και τώρα υπάρχουν, τρέχουν διαδικασίε κατά αυτή τη υπόθεση. Επίση, άλλο στόχο στρατηγικό είναι το να γίνουμε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να σχολιάσω επιδοκιμαστικά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Μαυροφούνιο καλωσορίζει τη στρατηγική αυτή, είναι ενθαρρυντική για την περιφέρεια και την περιοχή μα και δίνει ένα σαφέ μήνυμα για τι προοπτικές μα. Παρότι καλωσορίζουμε τις ενδεικτικές ημερομηνίε που αναφέρθηκαν, πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο στοιχείο της στρατηγικής είναι το μήνυμα που στέλνει ότι η πολιτική διεύνεση είναι ζωντανή. Φυσικά καλωσορίζουμε και το μήνυμα που προκύπτει από τη στρατηγική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση της αρχής της ε, ε, επιμέρους αξιολόγησης της πρόοδου της χώρας. Όσον αφορά την τρίτη μας προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική, οι καλές σχέσεις γειτονίας, το Μαυροβούνιο ήδη δρά ως κράτος μέλος που συμμερίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Συχνά έχουμε υποστηρίξει τις, τις γειτονικές μας χώρες, το Κωσυφοπαίδιο για παράδειγμα, ώστε να καλύψει τους όρους που απαιτούνται για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μας. Έτσι θα προσεγγίσουμε και τα άλλα ζητήματα με τους γειτονές μας ε, επικοδομητικά. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν πλέον προβλήματα. Ως απόδειξη της δέσμευσής μας για την περιφερειακή συνεργασία θα ήθελα να σας ανακοινώσω μια πρωτοβουλία της χώρας μου, την σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος βιώσιμων τεχνολογιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος του έργου αυτού είναι η εισαγωγή σύγχρονη θεραπεία για τον καρκίνο στου πολίτε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είχαμε καταπληκτική ανταπόκριση από του συναδέλφου μα στην περιοχή για την πρωτοβουλία αυτή. Αναμένουμε το μνημόνιο συνεργασία να υπογραφεί από του υπουργού ε, των συμμετόχων χωρών ε, στη Σύνοδο Κορυφή τη Σόφια το Μάιο φέτο. Κυρίε και κύριοι, η βασική αναπτυξιακή στόχη του Μαυροβουνίου μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι η σταθεροποίηση, η ανάπτυξη τη οικονομία μα και η πλήρη δέσμευση με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Το 2017 το ΑΕΠ μας ανήλθε κατά πάνω από 4%. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το κρατικό μας χρέος ε, το 2020 σε κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τη διαπραγματευτική διαδικασία, το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει μέχρι στιγμής 30 κεφάλαια. 30 κεφάλαια. Έχουμε κλείσει προσωρινά τρία κεφάλαια και έχουμε δεσμευτεί για να τηρήσουμε τα, benchmark, ε, τα ενδιάμεσα benchmark για τα κεφάλαια 23 και 24. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν ε, στη νέα φάση που πρέπει να περάσει το Μοντενέγρο, το και όλη η περιοχή. Εμείς στο Μαυροβούνιο πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα τρία κεφάλαια κατά τη Βουλγαρική Προεδρία. Όλα αυτά φυσικά βάσει των αποφάσεων που θα ληφθούν και εδώ εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν ικανοποιητικά για αμφότερες τις πλευρές. Επίσης, αναμένουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να κλείσουμε τις διαπραγματεύσει για κάποια από τα ανοιχτά κεφάλαια, όπω τα κεφάλαια 7 και 10. χάρη στο μεγαλύτερο ενθουσιασμό από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και εφόσον ε, υπάρξει και η ανταπόκριση από πλευρά του Μαυροβουνίου και ο ενθουσιασμό που χρειάζεται για να ανοίξουμε και τα επόμενα κεφάλαια, θα έχουμε αποκτήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την ορμή που χρειάζεται και εμεί πιστεύουμε ότι αυτό είναι δυνατόν. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μαζί να δώσουμε μια νέα όθηση στα κεφάλαια του τομέα του κράτους δικαίου, να καθορίσουμε τα κριτήρια αναφοράς για τα κεφάλαια 23 και 24. Είμαστε σίγουροι ότι φέτος θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα που θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες μας. Αλλά χρειαζόμαστε την υποστήριξη των θεσμικών οργάνων και των κρατομελών. μελών. Κυρίες και κύριοι, δεδομένου του γεγονότος ότι οι απόψεις διήστανται όσον αφορά την πρόοδο του Μαυροβουνίου, ειδικότερα για τα κεφάλαια που αφορούν το κράτος δικαίου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια συγκεκριμένα νούμερα. Και φυσικά θα σας δώσω και περισσότερες προφορές από το επιθυμείτε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Πρέπει να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Έχει δημιουργηθεί ήδη μια βάση στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ε, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ειδικότερα στους κόλπους του κρατικού μηχανισμού. Όλα αυτά είναι ορατά και στις δηλώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις δηλώσεις της κυβέρνησης μας. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ε, να υπάρχουν βιώσιμες συνθήκες. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να μπορούμε να επιτύχουμε νέα αποτελέσματα στο πλαίσιο που υπάρχει. Ε, όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση, έχουμε ολοκληρώσει τις βελτιώσεις ε, στο δικαστικό σύστημα που ξεκίνησαν με τις συνταγματικές τροποποίησεις του 2013. Αυτό είναι το τρίτο έτος που υλοποιούμε νομοθετικές καινοτομίες. Πολλές από αυτές ε, περιλαμβάνουν έναν ενίο μηχανισμό επιλογής για δικαστές και ε, κρατικούς αγγελείς, επαγγελματική αξιολόγηση, βάσει τι οποίε γίνονται και οι προαγωγές και επίδειξη ε, και λογοδοσία. Έχουν γίνει διάφορες μεταρρυθμίσεις, ε, μεταξύ των οποίων η σύσταση ενός ενιαίου εμπορικού δικαστηρίου, ενός κεντρικού οργανισμού ε, για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Έχουν, έχουμε δει ήδη τα αποτελέσματα πιο γρήγορες διεκπαιρώσεις των διαδικασιών και μείωση των ε, υποθέσεων που εκκρεμούσαν. Από την έναρξη του οργανισμού τον Ιανουάριο του 2016, 117 δημόσια λειτουργία έχουν παραιτηθεί βάσει γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων του οργανισμού. Όσον αφορά τα εισοδήματα, τα περισσοκά στοιχεία των αξιωματούχων, το 2017 όλες ε, οι δηλώσεις ε, εσόδων και ε, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων έχουν ελεγχθεί και σε 88 περιπτώσεις ε, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Τα γραφεία των εισαγγελέων ε, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή από τον Ιανουάριο του 2017 συστάθηκε το γραφείο του κριτικού εισαγγελέα που ασχολήθηκε με 1.615 υποθέσεις, από τις οποίες έχουν κλείσει 1.020. Στην καταπολέμηση της διαφθοράς το 2017 και μόνο έγιναν έρευνες για 76 φυσικά πρόσωπα και 17 νομικά πρόσωπα και μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών ε, κατηγορήθηκαν 18 ε, άτομα σε περιπτώσεις που αφορούν ε, διαφθορά εκδόθηκαν αποφάσεις για 24 άτομα εκ των οποίων 13 καταδίκες, 9 απαλλαγές και 20 περιπτώσεις ε, ε, κατηγορίας. Όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, το Γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα ξεκίνησε έρευνες κατά 68 ατόμων το 2017. Ε, διώχθηκαν 52 άτομα και κατηγορήθηκαν 19, καταδικάστηκαν 19 άτομα και εκδόθηκαν και απαλλαγές ε, για 21 άτομα. Επειδή είδαμε ότι έκανε προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυση των οικονομικών ερευνών, ήθελα να σας ενημερώσω ότι το 2017 οι οικονομικές έρευνες ε, αφορούσαν 19 υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος ε, για εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων. Όσον αφορά τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μόνο την τελευταία διετία μετά από πρόταση ε, του Γραφείου του Ειδικού Εισαγγελέα, το Ανώτο Δικαστήριο της Ποντγκόριτσα έδωσε εντολή για ασφαλιστικά μέτρα για κατάσχεση ιδιοκτησιών σε πάνω από 10 περιπτώσεις. Αυτό αφορούσε πάνω από 250.000 τετραγωνικά μέτρα ε, γραφείων ε, και κατοικίας. Έχουμε εξίσου καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις κατασχέσεις ιδιοκτησίας, διότι έχουμε κατασχέσει πολλές κατοικίες και πολλές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα γης, πολλά στρέμματα γης. Δεν θέλω να σπαταλήσω όλο το χρόνο σας αλλά είναι σημαντικό πιστεύω να σας ε, εκφράσω τη σαφή θέση της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου όσον αφορά τον τέταρτο πυλώνα του κράτους, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση τηρεί την αρχή των ανεξάρτητων μέσων ε, ενημέρωσης, της ελευθερίας έκφρασης και της προστασίας του κοινού και καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια ή δράση παρεμβολή ε, ε, στην εκδοτική δραστηριότητα ή στα μέσα μαζική ενημέρωση. Έχω επανειλημμένω δηλώσει ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά εκπροσώπου των μέσων ή περιφερειακών στοιχείων των μέσων είναι επίθεση προς τη δημοκρατία. Παραμένω ε, στη διάθεσή σα για να συζητήσουμε το θέμα αυτό εφόσον σας ενδιαφέρει. Τέλο, αγαπητοί συνάδελφοι, σα παρακαλώ επιτρέψτε μου να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα υιοθετήσουμε φέτος θα αναγνωρίσει την πρόοδο του Μαυροβουνίου και θα αποτελέσει μια επιπλέον δύναμη που θα οθήσει προς τα μπρος ε, την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια από τις σημαντικότερες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσετε και παραμένω στη διάθεση σας για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Mr. Deputy Prime Minister, thank you for your presentation and it seems like you are σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και φαίνεται ότι έχετε μπει στο σωστό δρόμο και τώρα θα αρχίσουμε το διάλογο με του ευρωβουλευτέ. Πρώτο ομιλητή είναι ο κύριος Τσάρλ Τάνοκ, που είναι ο μόνιμο εισηγητή τη ΑΦΕΤ για το Μαυροβούνιο. Κύριε Τάνοκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε αντιπρόεδρε τη κυβέρνηση, ε, νομίζω συναντηθήκαμε τελευταία φορά που ήμασταν στην Ποντγκόριτσα. Κάνατε μια... Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση αυτή. Το Μαυροβούνιο φαίνεται να κάνει τα σωστά πράγματα όσον αφορά την ιεράρχηση, το κράτο δικαίου, μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου και έρευνε ε, ακόμα και για υψηλά ειστάμενου υπαλλήλου στον αγώνα κατά τη διαφθορά μέσω του ρόλου σα ω Υπουργού δικαιοσύνη του Μαυροβουνίου. Αναμένουμε βεβαίως η Κομισιόν να προετοιμάσει έκθεση. Κάποια στιγμή ελπίζουμε τον Απρίλιο και έπειτα εγώ θα προετοιμάσω τη δική μου τελευταία έκθεση ως εισηγητής για το Μαυροβούνιο, αλλά πόσο μπορώ να δω μέχρι στιγμής και μετά από την επίσκεψή μου στην Ποτγκόριτσα, είστε στο σωστό δρόμο και είστε ο πρώτος υποψήφιος για ένταξη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοώ ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζαν Κλοντ πρόσφατα επισκέφθηκε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μετά από την δημοσίευση της ανανεωμένης στρατηγικής από πλευράς της Κομισιόν, που βέβαια ήταν ε, κάπως επιμαχό έγγραφο, γιατί είχε βάλει μια ε, διαφορετική ημερομηνία για το Μαυροβόνιο. Ελπίζω ότι η επίσκεψή του ήταν θετική. Ε, είχε μια επιτυχή σειρά συναντήσεων με εσά και διάφορα άλλα μέλη της κυβέρνησης και τώρα ευρύτερα, επειδή εσείς είστε μέλος της κυβέρνησης, πέρα από το ότι είστε Υπουργός Δικαιοσύνης, είστε και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κυβέρνησης σαφώς ε, προσλάβουμε στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου δύο τουλάχιστον οι περισσότεροι υποψήφοι υπάρχουν με τον, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργό Ζουκάνοβιτς και το Κοινοβούλιο θα στείλει μια ε, αποστολή παρακολούθησης των εκλογών. Ο Φάβιο Μάσιμο Καστάλντο, που είναι συνάδελφός μας σε αυτή την επιτροπή, θα, είναι, θα μετέχει σε αυτήν. Το άλλο θέμα είναι η ελευθεροτυπία. Υπάρχουν διάφορες δίκες που βρίσκονται υπό εξέλιξη Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εκείνη η δίκη εναντί δύο Ρώσων πολιτών που, που προσπάθησαν να στήσουν πραξικόπομα στη χώρα σας. Πολύ σημαντικό, ε, σημαντική υπόθεση δεδομένων των προβλημάτων που προέκυψαν μεταξύ της δικής μου χώρας, ε, των Ηνωμένων Βασιλείου και της Ρωσίας ε, με την απόπειρα και επιτυχία της δολοφονίας του κ. στο Σάλσμπουρι. από ό,τι φαίνεται η Ρωσία υποκινεί και παροτρύνει διάφορες ε, ενέργειες σε ξένες χώρες. Από φαίνεται τώρα έχει φυλακιστεί ο κ. Κνέσεβιτς. Εγώ τον συνάντησα στο Ποτκόριτσα. Ήταν αρκετά γεννής και προσβλητική. Μπορώ να πω ότι δεν θα λυπηθώ αν πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Αλλά βέβαια δεν θα πρέπει να είναι κανείς πέρα από τον νόμο εάν διαπράττει ποινικά δικήματα. Και θα προετοιμάσουμε και τη σχετική έκθεση ε, μέσα στο χρόνο. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερλε τώρα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη, χαρά μου που να σας ε, βλέπω και πάλι. Ε, μπόρεσα να επισκεφθώ τη χώρα σας ε, πανελειμμένα τον τελευταίο καιρό και κάθε φορά διαπιστώνω την πρόοδο. Και δεν το λέω για να σας κολακέψω, αλλά ε, ειλικρινά το λέω, είμαι πολύ ικανοποιημένο και ευτυχής που το Μαυροβούνιο έχει βάλει πλώρη για την ένταξη. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια σημεία. Εσείς αναφέρατε πολλά από αυτά που ήθελα ήδη να πω. Ε, είναι σαφές ότι το Μαυροβούνιο γνωρίζει ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Συμφωνούμε επίσης ε, για το ότι η νέα στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια δίνει μια νέα όθηση στη διαδικασία. Είναι σημαντικό να μην επικρατήσει κόποση, ε, να διατηρηθεί ζωντανή η βούληση και ε, είμαι πεπισμένος ότι εσείς ε, όπως και εγώ θα θέλαμε η διάσκεψη κορυφής της Σόφιας θα αποτελέσει μια προσθεθέμενη αξία. Επίσης ήθελα να εκφράσω την χαρά μου για τα όσα είπατε για το καρκίνο γιατί εγώ είμαι πρόεδρος της ομάδας της Ένωσης για τον αγώνα κατά του καρκίνου. Και Ελπίζουμε και πάλι ότι η διάσκεψη κορυφή τη Όφιας που θα ασχοληθεί με το θέμα θα εκπονηθεί εκεί και έκθεση σε σχέση με το θέμα αυτό και ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα ε, είναι επιτυχής αυτή η προσπάθεια. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχηθώ σε εσά και στη χώρα σας ε, μετά από τις εκλογές. Ε, να συνεχίσει να προχωρά σε αυτή τη διαδικασία την προταξιακή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πέτρελε. Ο κύριο Πίτσουλα. Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη, μεγάλη μας χαρά που σας βλέπουμε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας. Εγώ δεν θα σας υποβάλω ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα μόνο να μοιραστώ μαζί σας ένα προβληματισμό σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Μαυροβούνιο, που είναι στη πρόθυρα της ένταξης. Είναι σαφές ότι ζωβούν διάφορες κρίσεις στην ε, χώρα σας, στα άμεσα σύνορα, όπως ε, επίσης και στο εσωτερικό της χώρας. Και για αυτόν τον λόγο για Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σας πω ότι ζει το ίδιο και γι' αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και κατά καλά νέα από το Μαυροβούνιο. Πιστεύω πως οι Βρυξέλλες ε, θα πρέπει να τιμήσουν το λόγο τους Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο στην επίλυση των ιστορικών του προβλημάτων θα πρέπει να βασιστεί στην διεύρυνση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα Βαλκάνια να ε, είναι και πάλι μια περιοχή που θα αρχίσει να ανησυχεί την Ευρώπη. Ήδη σοβούν διάφορε κρίσει, η οικονομική, η προσφυγική. Δεν χρειάζεται ακόμα μια κρίση στα Βαλκάνια. Νομίζω λοιπόν πως το Μαυροβούνιο δεν έχει τα προβλήματα που, τα οποία υποφέρουν άλλες χώρες των Βαλκανίων ε, στη φάση της διαπραγμάτευσης και αυτό το λέω έχοντας γνώση του θέματος γιατί εγώ παρακολουθώ τις σχέσεις με τη Βοσνία Ζεγοβίνη και το Κωσυφοπαίδιο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, κερδίσουν αυτοί που προχωρούν περισσότερο στο δρόμο της ένταξης. Δεν μπορούμε όλους να τους αντιμετωπίζουμε ομοιόμορφα. Και θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάποια πράγματα ε, και αυτό σας το ρωτώ ως Κροάτης με την εμπειρία που έχω. Βλέπουμε ότι στη χώρα σας υπάρχουν κόμματα πολύ πολλωμένα. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι στην πρόοδο, γιατί το Κοινοβούλιο ε, πρέπει ακόμα να εγκρίνει πολύ σημαντικές νομοθεσίες που είναι θεμελιώδεις για την πρόοδο προς τη διεύρυνση. Θα γίνουν προεδρικές εκλογές ε, και θα μπορούσα να έρθω στο Μαυροβούνιο ως παρατηρητής. Και ακριβώς θα ήθελα να γνωρίζω τι θα κάνετε για να βγείτε από αυτήν την ε, κατάσταση πώλησης που όπως είπα μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι. Δηλαδή μιλώ για τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας και όχι τόσο για εμπόδια στην ε, ενταξιακή πορεία. Ευχαριστώ κύριος Μέζεριτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξοχότατε την πρόεδρε τη κυβέρνηση, κύριε Πρέσβη, σα καλωσορίζω και εγώ στην συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η δική μου πολιτική ομάδα την χάνει να είναι από εκείνε που ανέκαθεν ήταν αναφαδόν υπέρ της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Και σήμερα πιστεύουμε, αλλά και στο παρελθόν φρονούσαμε ότι η δέσμευση της Θεσσαλονίκης το 2003 θα πρέπει να τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επανέλθουμε με τη νέα στρατηγική στις παλιές αυτές πολιτικές. Έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι έχουν επιδεινωθεί κάποια πράγματα. Ε, αυτή η πορεία είναι διπλής κατεύθυνσης. Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποιες προσπάθειες, αλλά και οι υποψήφιες χώρες από κοινού. Με βάση αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας αναφέρω δύο πράγματα για τα οποία ανησυχεί ιδιαίτερα η δική μας πολιτική ομάδα. Και τα δύο είναι σημαντικά σε σχέση με τη χρηστή διακυβέρνηση και γενικότερα τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζουμε όλες τις βελτιώσεις που έχετε κάνει, αλλά θα θέλαμε να δούμε ή δυνατόν περισσότερες βελτιώσεις στην πρόσβαση στη δημόσια ενημέρωση. Ανησυχούμε για κάποια από τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ε, τα μεγάλα έργα υποδομών και φυσικά η ομάδα των Πρασίνων ενδιαφέρεται παγίως για έργα που κατασκευάζονται ε, σε προστατευόμενες περιοχές, υδροελεκτρικά ε, φράγματα δηλαδή και ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Τα γνωρίζετε όλα αυτά, αλλά ε, θα μας ενδιέφερε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού. Δεύτερον, χαίρομαι πάρα πολύ για την αναφορά σας στην ελευθεροτυπία. Διαπιστώνουμε κι εμείς ότι η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου είναι προσιλωμένη στην ελευθεροτυπία υπό όλες τις έννοιες και συμφωνούμε, αλλά ανησυχούμε παρόλα αυτά για πρόσφατες επιθέσεις, πιέσεις, απόπειρες ε, εκφοβισμού ε, με απειλές και κατά της σωματικής ακαιρεότητας. Ε, εσείς πώς μπορείτε να πιέσετε και να τελειώσει η υπόθεση του Ντούσκο 14 χρόνια κρεμεί αυτή η δολοφονία που είναι κάπως υπερβολικό ακόμα και για βαλκανικούς όρους. Και επίσης ανησυχούμε ε, με τις διάφορες συκοφαντικές ε, δυσφημίσεις κατά δημοσιογράφων όπως είναι η περίπτωση Μαρτίνοβης ε, που δεν θεωρούν πολύ ότι έχει γίνει δίκαιη έτσι, δικαστική διαδικασία. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστάλτο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ σας, σας ευχαριστώ εξοχότατε κυρία την Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Πρέσβη, κυρίως για αυτή την πολύ ε, σημαντική ενημέρωση που μας δίνει την κατάσταση προόδου όσον αφορά τις προσπάθειες, τις σημαντικές που κάνει το Μαυροβούνιο. Όπως είπε πολύ καλά ο συνάδελφος Τσάρλς Σάνο που γνωρίζει βαθιά τη χώρα σας αυτή τη στιγμή, είναι η ε, πρωτοπόρα χώρα στην ε, διαδικασία την πεντεξική και είμαι ευτυχής που η σημερινή βουλγαρική προεδρία έδωσε έμφαση στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων που πρέπει να μπουν μέσα στην Ένωση. Ιδιαίτερα διαπίστωσα με χαρά τις προσπάθειες που γίνονται στο πεδίο της δικαιοσύνης, ε, στα όσα μας είπατε για τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς εξάλλου. Για πρώτη φορά εγώ επισκέφθηκα τη χώρα σας πέρυσι για ένα σεμινάριο στην Ράσπα, τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, και μάλιστα ήρθα με άλλους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με πολλές αντιπροσωπείες ε, στις, ε, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Από αυτή την άποψη λοιπόν συμμερίζομαι ε, την ενθάρρυνση που σας έδωσαν οι περισσότεροι συνάδελφοι και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να προχωρήσετε και στα υπόλοιπα κεφάλαια, να μπορέσετε να κλείσετε και αυτά που είναι ακόμα ανοιχτά, γιατί σας θεωρούμε κάπως το υπόδειγμα και την ε, το κίνητρο και για τις υπόλοιπες ε, γειτονικέ σας χώρες. Θα ήθελα μάλιστα να σας ρωτήσω, να κάνω μια παρατήρηση, γιατί πολλά ζητήματα τα έθιξαν οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν. Ένα πρόβλημα που εν μέρει έχουμε κοινό και είναι οι ξένοι μαχητές από τη Μέση Ανατολή, ο κύριος από τη Συρία. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πλήττει και τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν έχουμε ακόμα ακριβεί στατιστικέ για το ποιο ποσοστό έχει έρθει στο Μαυροβούνιο όμως μπορεί να κάνουν όχι μόνο τροποκρατικέ απόπειρε, αλλά μπορεί να συμβάλλουν και στη ριζοσπαστικοποίηση και στην αύξηση του θρησκευτικού εξτρεμισμού και βέβαια σημαίνει μεγαλύτερο κινδύνους λόγω των ε, τις εμπειρίες τους που επέκτησαν στον πόλεμο. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε λοιπόν ποια συγκεκριμένα μέτρα έχετε λάβει εάν έχετε εστιάσει σε σκληρές πολιτικές, δηλαδή στο να ε, οξύνεται κάπως ή τα μέτρα στο ποινικό πεδίο ή αν έχετε εστιάσει στην ένταξη των ξένων αυτομαχητών στην κοινωνία πόσο επηρεάζει αυτό το φαινόμενο δηλαδή την επικρατεία σας και Τέλος, να σας θαρρύνω και πάλι να συνεχίσετε σε αυτήν την ε, αγαστή πορεία. Ελπίζουμε ότι το κλίμα αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση θα βρει το δρόμο στον κοινοβουλευτικό και θα εγκαταλειφθεί το σαμποτάζ γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι θετικό για να προχωρήσετε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και ελπίζουμε ότι γρήγορα θα μπείτε και εσείς στη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ. Πετήρ. Κυρία Πετήρ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε την Πρόεδρε της Κυβέρνησης. Κύριε Πρέσβη. τέλη Ιανουαρίου τα μέσα ενημέρωσης μας ενημέρωσαν για την παραβίαση των δικαιωμάτων των Κροατών στο μοτοσυκό. Πρόκειται για ένα γνωστό πρόβλημα που υπήρχε με την Κροατία γιατί η Κροατία ζήτησε να εγγραφεί ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της Κροατίας, Κροατική, στην ε, UNESCO. Πρόκειται για ναυτικούς που έχουν πολύ παλιά παράδοση κροατική, πάρα πολύ παλιά. και παρόλο που είναι κροατική αυτή η παράδοση, δεν μας ζητήσατε τη γνώμη μας, εμάς. Ε, οι μειονότητες έχουν δικαιώματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάζονται τα δικαιώματα της ε, κροατικής μειονότητας, του κροατικού πληθυσμού. Τι προτίθεται να κάνει το Μαυροβούνιο. Θα ζητήσει μαζί με την Κροατία ε, να ενταχθεί στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά ως κροατική κληρονομιά και θα αλλάξετε τακτική απέναντι στους Κροάτες. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ο κύριος Μποστινάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, πέρυσι υπήρξε αυτό το περίφημο πραξικόπημα ή απόπειρα πραξικοπήματος ε, μια συνωμοσία διαφόρων φορέων κρατικών και μη κρατικών. Τι θα μπορούσατε σήμερα να μας πείτε για όλα αυτά, χωρίς να αποκαλύψετε καμιά απόρριτη πληροφορία. Πώς έχετε μάθει περισσότερα σε σχέση και σύγκριση με την προηγούμενη ενημέρωση. Και τι κρύβεται πίσω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Και δεύτερον, το Μαυροβόνιο πώς βλέπει σήμερα τους παράγοντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν πάρα πολύ να εμπλακούν στα Δυτικά Βαλκάνια. Και τι συμβουλή θα δίνατε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει αυτό το κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. So, easy Εύκολες ερωτήσεις για τον κύριο Πασίν. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, έχετε το λόγο. Well, Ωραία, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα αξιότιμα μέλη που εκδήλωσαν ε, το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο του Μαυροβουνίου καθώς ε, προχωρά σε αυτό το δρόμο για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια ευκαιρία για μένα να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου. Κύριε Τάνοκ, λυπάμαι ειλικρινά που ακούω ότι αυτή είναι η τελευταία σας έκθεση για το Μαυροβούνιο. Αυτό διότι έχετε δείξει ιδιαίτερο επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα. Αυτή είναι και η άποψη των πολιτών του Μαυροβουνίου και δράτω με τις ευκαιρίες για να σε ευχαριστήσω. Ως ε, βουλευτής εδώ και χρόνια επισημαίνεται ότι φυσικά υπάρχουν δεσμεύσεις από πλευράς του Μαυροβουνίου όσον αφορά την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες πτυχές ε, είναι επίμαχες. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τις επιμαχίες πτυχές, διότι η δέσμευσή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προσχώρησή μας είναι πλήρης. Αυτή φυσικά βασίζεται στη δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων και ολοκλήρης της κοινωνίας, διότι ένταξη αφορά, είναι κάτι που αφορά την κοινωνία στο συνολό της, όχι μόνο τους θεσμούς της. Θέλουμε λοιπόν εμείς ε, να προχωρήσουμε σε ποιοτικές μεταρρυθμίσεις και να γίνουμε μείζον εταίρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την άψη. Η φετινή χρονιά ενέχει πολλές προκλήσεις στις οποίες θα ανταποκριθούμε με τη δημοκρατική οριμότητα που θα αναγνωρίσουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είπατε. Θα έχουμε τις προεδρικές εκλογές ε, στα μέσα Απριλίου, τις οποίες θα ακολουθήσουν κοινοβουλευτικές εκλογές σε 12 περιφέρειες. Η δημοκρατία μας ε, με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί. Οι εκλογές αυτές θα δώσουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή του Μαυροβουνίου. Το Μαυροβουνίο φυσικά παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ε, μιας ε, συγκεκριμένης δύναμης η οποία είναι δυσαρεστημένη με την ιδέα της ένταξης του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πορεία του Μαυροβουνίου για ένταξη στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο δεν έχει σκοπό να βλάψει κάποιον, ούτε είναι κάτι που κάνουμε κατά κάποιου. Σκοπό έχει την ενίσχυση του συνόλου της κοινωνίας μας. Αν σκεφτείτε όλες τις προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι στιγμής, έχουμε ε, καλύψει τις απαιτήσει με δημοκρατική οριμότητα. Οι θεσμοί μας έχουν καταφέρει να βρουν απαντήσεις και το δικαστικό σώμα επίσης θα βρει κάποιες απαντήσεις. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται δίκες για τρομοκρατικές πράξεις ε, και εγκληματικές οργανώσεις. Κύριε Πέτρελε, ευχαριστώ που αναγνωρίζετε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ειδικότερα γνωρίζοντα ότι η ενθάρρυνση αυτή προέρχεται από μια φιλική χώρα προς εμάς όπως η Σλοβενία. Όπως έχετε ακούσει ήδη, ε, φέτος προγραμματίζουμε να ανοίξουμε τα υπόλοιπα κεφάλαια ε, που αφορούν την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κλείσουμε και κάποια κεφάλαια. Και ένα πράγμα είναι βέβαιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι διαπραγματεύσεις που αφορούν 20, ε, τα, τα κεφάλαια 23 και 24 είναι πολύ σημαντικές. Ειδικότερα η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένας από τους πυλώνες ε, της προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά με τρόπο υπεύθυνο και όρεμο. Φυσικά πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όταν θεσπίσει κανείς συστήσει κάποια, ε, κάποια όργανα, κάποια θεσμικά όργανα, πρέπει να του δώσει και λίγο χρόνο για να φέρουν αποτελέσματα. Και εγώ είμαι βέβαιο ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα δούμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ επίση που αναγνωρίζετε τι προσπαθίε μα όσον αφορά την περιφερειακή προσέγγιση των βιώσιμων τεχνολογιών και όπως αναφέρθηκε θα γίνουν και περισσότερες συνομιλίες για το θέμα αυτό στη Συνοδοκορυφή της Σόφιας. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε για την πολύ σαφή σας δήλωση όσον αφορά την ουσία της εξωτερικής πολιτικής του Μαυροβουνίου. Ειδικότερα όσον αφορά τις σχέσεις Μαυροβουνίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, η επιθυμία μας να συμβάλλει το Μαυροβούνιο πλήρω στη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, το Μαυροβούνιο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Σταθερότητα αντί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεδομένη της γεωγραφικής θέσης του Μαυροβουνίου να είμαστε παραγόντας σταθεροποίησης. Και ευχαριστούμε επαναγνώριση ότι δεν υπάρχουν εκρεμή ζητήματα από αυτή την άποψη όσον αφορά το Μαυροβούνιο. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το τεράστιο πολιτικό μας κεφάλαιο. Δεδομένου ότι στη σκοτεινή δεκαετία του 90 κατά τη διάρκεια των πολέμων στα Βαλκάνια δεν υπήρξαν σειράξει μεταξύ εθνοτήτων στο Μαυροβούνιο. Καταφέραμε να διατηρήσουμε εκείνη την εποχή την ειρήνη στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο σήμερα το Μαυροβούνιο έχει πολύ καλές σχέσεις με τις γειτονικές ε, χώρες, όλες τις γειτονικές χώρες και μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν. Όλα τα Δυτικά Βαλκάνια φιλοδοξούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Χάν και από τον κύριο Γιούνκερ, τα εκκρεμή ζητήματα που απομένουν μεταξύ αυτών των ε, επίδοξων μελών θα πρέπει να επιληθούν. Αναφέρατε επίσης τις ε, πολλωμένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών κομμάτων του Μαυροβουνίου. Αυτός είναι ένας περιορισμός που επιβάλλεται στην κουλτούρα του διαλόγου που υπονομεύτηκε πέρυσι μεταξύ άλλων λόγω του ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Κοινοβουλίου μποϊκόταραν τις συνομιλίες ε, και λόγω κάποιας μορφής ρητορική που ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες, ειδικότερα από ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο εξέφερε ε, σαφή αποδοκιμασία όσον αφορά την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλω να δηλώσω σαφώς ότι εμείς θα απαντήσουμε, μάλλον οι πολίτες θα απαντήσουν σε όλα αυτά τα διλήμματα. Και πολύ σύντομα μάλιστα. Πολύ σύντομα θα έχουμε προεδρικές εκλογές και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ε, εκλογές ε, σε 12 αυτοδιοικούμενες ε, περιοχές και εκεί θα καταστεί σαφές ποια είναι η επιθυμία του λαού. Φωνή λαού, φωνή Θεού, Vox Populi, Vox Dei. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι όλοι οι παράγοντες της πολιτικής κοινής και όλοι οι πολιτικοί εταίροι θα συνταχθούν πίσω από ένα κοινό συμφέρον που είναι μια δυναμική κοινωνική και οικονομική πρόοδος του Μαυροβουνίου. Κυρία Μέσερετς, Ένα, αυτό που αναφέρατε είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, η ελεύθερη πρόσβαση στις ε, πληροφορίες. Ε, και έτσι αυτό το δικαίωμα πρέπει να το ενισχύσουμε εντός της Ευρώπης. Ε, είναι κομμάτι όλο αυτό της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ελευθερίας ε, των πολιτών και, γιατί ξέρετε μόνο οι πολίτες που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ελεύθερα μπορούν να έχουν την ελευθερία έκφρασης της απόψής τους. Είναι ενδιαφέρον ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο δίστασε για πολύ καιρό να υιοθετήσει μια τέτοια προσέγγιση ελεύθερη πρόσβαση τη πληροφορία και μόνο μόλις πριν από λίγα χρόνια και μάλιστα είναι σωστά θα έλεγα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε αυτό το δικαίωμα ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρωπίνα δικαιώματα. Φυσικά οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, σε πληροφορίες όσον αφορά μεγάλα κατασκευαστικά έργα, έργα υποδομής, όσον αφορά επίσης οικολογικά ζητήματα και φυσικά το Μαυροβούνιο το γνωρίζει. Εμείς ε, εμένουμε στην ελευθερία έκφρασης σύμφωνα με τα όσα είπατε και εσείς. Είναι σαφές ότι η ελευθερία έκφρασης έχει μια βασική πτυχή την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Και όπως είπα, οποιαδήποτε επίθεση κατά το ΜΟΜΟΕ, όπως ε, απειλές, επιθέσεις προς δημοσιογράφους, ε, καταστροφή περιουσιακών στοιχείων των μέσων μαζική ενημέρωση αποτελεί ταυτόχρονα επίθεση κατά της δημοκρατίας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου συνέστησε μία επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφους, με στόχο τη διερεύνηση την ε, διαγωγή των κρατικών θεσμών από αυτή την άποψη. Και εδώ έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, διότι η κυβέρνηση δέχτηκε όλες τις συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή αυτή. Η κυβέρνηση λοιπόν υιοθέτησε όλες τις συστάσεις. Και ενθάρρυνε δημόσια την Επιτροπή αυτή να συνεχίσει το έργο της. Εκχωρώντας και τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να συνεχίσει τις εργασίες της. Αναμένουμε ότι η αστυνομία, η κρατική εισαγγελία και άλλοι κρατικοί θεσμοί που εμπλέκονται στο θέματα αυτά θα μας διατηρούν ενήμερους όσον αφορά την προσέγγιση της κυβέρνησης στα θέματα αυτά. Φυσικά, όταν μιλάμε για αυτή την έρευνα, αναφερόμαστε και στην πολύ δύσκολη περίπτωση της δολοφονίας του Ντοσκο Ιωβάνοβιτς. Ένα καθήκον της Επιτροπής είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την υπόθεση αυτή μετά από την τραγική η ε, δολοφονία αυτή. Φυσικά αυτό που είπαμε όσον αφορά την εστίαση της Βουλγαρικής Προεδρίας στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια ή όπως εμάς ε, ε, εμείς προτιμάμε να λέμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Βουλγαρική Προεδρία που υιοθέτησε τέτοια θέση. Επίσης μιλήσατε για τους αλλοδαπούς μαχητές που επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή. Μας ρωτήσατε πώς ε, ασχολούμαστε με το πρόβλημα αυτό, τι κάνουμε. Είμαστε επεπισμένοι ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιληθεί με πολυτομιακό τρόπο. Γιατί, διότι δεν αρκεί να το αντιμετωπίσουμε μόνο ποινικά ή νομικά. Εντάξει, να αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα, έχουμε αναγνωρίσει ότι η συμμετοχή ε, σε ε, μάχες ως αλλοδαπός μαχητής είναι εγκληματική πράξη, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα όπως επανεκπαίδευση, παιδεία, καλή συνεργασία μεταξύ του κράτους και της θρησκευτική κοινότητα, ώστε να προλαμβάνουμε πιθανή ριζοσπαστικοποίηση στο μέλλον αλλοδαπών μαχητών. Ε, και φυσικά είναι σημαντικό να υπάρχει καλή συνεργασία με τις άλλες χώρες. Διότι το πρόβλημα αυτό φυσικά δεν είναι μόνο χώριο, είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια διαδραστική προσέγγιση εδώ για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής το Μαυροβούνιο δεν έχει αναγνωριστεί ως ε, προβληματική χώρα, ως χώρα όπου το πρόβλημα αυτό κλιμακώνεται σε ανησυχητικό βαθμό. Είχαμε δύο υποθέσεις ε, αλλοδαπών μαχητών. Αυτό όμως δεν σημαίνει παρά το ότι πρέπει να συνεχίσουμε τα προληπτικά μέτρα γνωρίζοντας ότι η καταστολή δεν είναι παρά αντίδραση συνήθως παρότι ενίοτε η καταστολή μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά. Μιλήσατε για την κροατική μειονότητα και τις παραβέσεις των δικαιωμάτων ε, στην ΠΟΚΑ. Διαφωνώ με τα όσα είπατε. Διότι τα μέλη της κροατικής ε, κοινότητας ε, χαίρουν σεβασμού και αναγνωρίζονται. η κρατική μειονότητα εκπροσωπείται και στο Κοινοβούλιο. Και αυτό είμαι βέβαιο δεν θα συνέβαινε αν τα μέλη της κοινότητα αυτή ε, αισθάνονταν απειλή ή ότι κινδυνεύουν στο Μαυροβούνιο. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας ε, όλα τα μέλη όλων των μειονοτήτων να αισθάνονται άνετα στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο δεν είναι κράτος μιας εθνότητας, είναι ένα κράτος πολιτών. Και όταν τίθεται το ερώτημα της υποψηφιότητας που έκανε που θα πρέπει να αναγνωριστεί από την ε, UNESCO, μάλιστα, πρόκειται πιστεύω για μια πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να φέρει πιο κοντά όλους τους πολίτες του Μαυροβουνίου, ειδικότερα εκείνους που έχουν ιδιαίτερη θέση στην ΠΟΚΑ, όπως ε, η κροατική ε, εθνική μειονότητα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να πω ότι οποιοδήποτε πολιτιστικό προνόμιο του Μαυροβουνίου σύμφωνα με το Σύνταγμά μας είναι ένα προνόμιο που ανήκει σε όλες τις κοινότητες και όχι μόνο σε μία και όχι σε άλλες. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι το Μαυροβούνιο είναι ένα κράτος πολιτών και όχι εθνοτικών ομάδων. Αν ε, ψάξετε να δείτε το σύνταγμα, ε, τα συντάγματα των χωρών της περιοχής, θα παρατηρήσετε ότι το σύνταγμα αναφέρεται κυρίως ε, σε έθνη των κρατών αυτών. Ενώ αυτό συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη της περιοχής, ενώ στο Μαυροβούνιο ε, αναφερόμαστε ως, στο Σύνταγμά μας ως χώρα πολιτών. Φυσικά συμφωνώ μαζί σας, η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το Μαυροβούνιο. Και θα συζητήσουμε την πρωτοβουλία αυτή με τους εκπροσώπους της κρατικής μειονότητας στο Μαυροβούνιο. Θα γίνουν φυσικά συνομιλίες και γίνονται ήδη συνομιλίες με το Υπουργείο Πολιτιστικής Δημιουργίας και το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Κροατίας. Και τέλος, ε, ο κ. Μποστινάρο ρώτησε κάτι σχετικό με το υπόβαθρο, το πλαίσιο, τη λογική που διέπει την υπόθεση που περιγράφεται ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ε, δημιουργίας εγκληματικής ομάδας. Εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός όταν συζητάω ε, δικαστικές υποθέσεις που τρέχουν. Ε, το δικαστικό σώμα θα έπρεπε να δίνει τις σχετικές απαντήσεις. Ωστόσο, εμείς στην κυβέρνηση δεν έχουμε καμία εμφιβολία. ότι πρόκειται για ε, αναρμόζουσα ε, ξένη παρεμβολή σε εγχώρια ζητήματα και ο λόγος ήταν πρώτα απ' όλα να παρεμποδιστεί η προσχώρηση του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, το αυτή συγκεκριμένη δύναμη είδε την προσχώρηση αυτή ως παρεμπόδιση των δικών του εθνικών συμφερόντων. Ενώ αυτό δεν συνέβαινε σε καμία περίπτωση το Μαυροβούνιο, επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις με όλους συμπεριλαμβανομένες και εκείνης της συγκεκριμένης χώρας, αλλά οι πολίτες του Μαυροβουνίου και μόνο θα είναι αυτοί που θα αποφασίζουν για το μέλλον του Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αν υπομονούμε να συνεχιστεί στο μέλλον η συνεργασία μας, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα δύο λεπτών. Κατσάρων λεπτών ε, είναι εδώ η κυρία Φώτηκα και θα γίνει η συζήτηση με τον, κύριο, με τον Επίτροπο τον κύριο Χάν και